αφορά τους διορισμούς στις κοινοβουλευτικέ επιτροπές. Τα σχετικά στοιχεία μπορεί να δείτε στα πρακτικά της συνεδρίασής μας και θεωρώ ότι εγκρίνονται